Bien, mes chers collègues. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Γκρέλστα και ο υποφαινόμενος θα προεδρεύσουμε τη κοινή αυτή συνεδρίασης. Πώς θα εργαστούμε τώρα, σε δύο τμήματα. καταλήξουμε δηλαδή και στο γενικό μας συμπέρασμα από τις 10 και μισή καταρχάς μέχρι τις 10 50 11 παρα 5, θα έχουμε μια παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 20 λεπτά και 20 ακόμα λεπτά στη συνέχεια με τη μέθοδο Catch the Eye για ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στη συνέχεια 5 λεπτά για να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα τις έχουν υποβληθεί Ερωτήσεις, όπως σας είπα, θα πρέπει να υποβληθούν σε ένα διάστημα 15 λεπτών και έπειτα θα ακούσουμε άλλη μια παρουσίαση κατά 20 λεπτά από τη Γενική Διεύθυνση Budget και έπειτα πάλι με τη μέθοδο Catch the Eye για 15 λεπτά θα μπορέσει να υποβάλλεται ερωτήσεις και στη συνέχεια θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συνέχεια θα ακούσουμε και κάποια συμπεράσματα, θα δούμε ποια διδάγματα θα μπορέσουμε να αντλήσουμε και ο κύριος Άσουαρθ και η κυρία Γκρέσλε θα μας διαφωτίσουν περισσότερο για τα συμπεράσματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρήσουμε το χρόνο αγόρευσης. Και εγώ με την κυρία Γκρέσλερ μπορούμε επίσης να σας δώσουμε και τη δυνατότητα πριν τις 31 Ιανουαρίου να υποβάλλετε ακόμα και γραπτά ερωτήσεις, αν δεν καταφέρετε να τις υποβάλλετε σήμερα προφορικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα για 8 ακριβώς σημεία που έχουν να κάνουν με κάποιες βασικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με το δημοσιονομικό κανονισμό και, τους προτινόμενους σε αυτόν, και τις προτινόμενες σε τροποποίησεις. Ο Βρατιμίρ Μάνκα από τους σοσιαλιστές, ο Λες Μιαλή από, το, την Άλντε, από την Κουέ η κυρία Ριάντα, ο Σερεβέρ, ο, ο Ίντρεκ Τάραντ, από το ΕΣΥΑΡ, Πετρή Αλβάμα από το ΕΛΚΑ, από τους σοσιαλιστές Νέσσα Γιάννα Σέντερ, από το ΑΛΔΕ, ο ίδιος και ο δισηγητής, και για τους πρασίνους Μπαρτ Στάισε. Οι Άγκρι, οι Ρέτζι, οι Έμπλη, οι Τραν, οι Ήτρε, οι Ντεβ, οι Λίμπε, οι Άφετ θα υποβάλουν γνωμοδοτήσει και έχουν ενημερωθεί για τη σημερινή παρουσίαση. Υπάρχει μάλιστα και ένα μνημόνιο συνεννόηση με πέντε από τι συνδεδεμένε αυτέ επιτροπέ, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού και εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των ε, Πρόεδρων των Επιτροπών στις 12 Ιανουαρίου και στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής Έχουμε, επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος για να εγκρίνουμε στις 11 Μαΐου το σχέδιο αυτοέκθεσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Μάρτιο θα έχουμε πάλι μια κοινή συνεδρίαση, 30 Μαΐου μάλιστα, κοινή συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής Προπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Κυρία Πρόεδρε, εκπροσωπώντας εσείς την ε, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω ευθύ αμέσω την παρουσίαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Θα ήθελα να τηρήσω λοιπόν τον χρόνο που μα δώσατε εσεί, κύριε Πρόεδρε. Η παρουσίαση σήμερα το πρωί θα επικεντρωθεί σε κάποια βασικά σημεία της τροποποίησης που προτείνουμε. Θα δούμε καταρχάς ποιες είναι οι δυνατότητες απλούστευσης που προβλέπονται για τους δικαιούχους, το νέο σύστημα ελέγχων, το νέο σύστημα λειτουργίας της χρηματοδότησης. Θα επικεντρωθούμε επίσης στον τρόπο εκτέλεσης του προπολογισμού, ευθυγράμμιση της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων και μεγαλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα. Α ξεκινήσουμε καταρχά με το σύστημα πλούστευση για του δικαιούχου, για του αποδέκτε. Γνωρίζετε ότι ε, αυτό ήταν από τα βασικά αιτήματα της δημόσιας διαβούλευσης. Πάρα πολλοί μας είπαν ότι έπρεπε να πλουστευτεί το σύστημα των κοινοτικών κονδυλίων για τους ίδιους τους δικαιούχους, για τους ίδιους αποδέκτες. Θέλαμε να έχουμε πιο απλούς κανόνες, γιατί είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους και των σφαλμάτων όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τις διοικητικές αρχές. Επικεντρωθήκαν λοιπόν στο ζήτημα της απλούστευσης από την αρχή της εφαρμογής μέχρι την καταβολή των τελευταίων ποσών, χρήση των κονδυλίων, ε, καταβολή πληρωμών και ex post έλεγχη και παληθεύσεις. Μας ε, ενδιαφέρουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για την ε, πληρωμή των κονδυλίων αυτών. Θα αναφερθούμε επίσης στην κατάργηση της αρχής της μη αποκόμισης του κέρδους Ξέρετε επίσης ότι όσον αφορά τις επιλογές ε, για τις απλουστευμένες μάλλον επιλογές για την παρουσίαση των δαπανών και εδώ θέλουμε μεγαλύτερη απλούστευση γιατί δεν θέλουμε υποβολή εκθέσεων που έχει να κάνει μόνο με το κόστος, μόνο με τις εισρωές αλλά και υποβολή εκθέσεων που να έχουν να κάνουν κυρίως με τα αποτελέσματα και δεν θέλουμε αναγκαστικά να έχουμε στη συνέχεια ex post ελέγχους όσον αφορά το ζήτημα αυτό των δαπανών. Καταλαβαίνετε ότι οι προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτόματα δεν, αυξάνουν σε, δεν καμία περίπτωση τις δαπάνες. Ας δούμε τώρα όλες αυτές τις αλλαγές μία προς μία, πολύ συγκεκριμένα. Τι κάναμε καταρχάς για το στάδιο της εκτέλεσης, προκειμένου να πλουστευτούν εδώ πέρα τα πράγματα για τους δυνητικούς ε, ε, συμμετέχοντες. Είπαμε καταρχάς ότι ε, για επιδοτήσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω των 750.000 ευρώ. Δεν θα προβλέπονται εδώ πέρα συγκεκριμένες απαιτήσει και το ίδιο θα ισχύει και για τις λειτουργικές επιδοτήσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Αν υπάρχει έλεγχος ο οποίος απαιτείται από τις εθνικές αρχές, τότε θα μπορεί να λαμβάνει η χώρα. Δεν θέλουμε όμως εμείς να επιβάλλουμε εκ των προτέρων ελέγχους και παληθεύσει. Θα το κάνουμε αυτό μόνο αν έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό που να υπερβαίνει το κατόφλι το οποίο σας παρουσίασα. Δεν θα προβλέπετε λοιπόν κάποιος έλεγχος, ιδίως για τους δικαιούς εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν αν θα λάβουν τελικά επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι έλεγχοι για την ε, μη σωρευτική αρχή πλέον καταργούνται. Θεωρήσαμε ότι δεν υπήρχε λόγος για αυτές τις κατηγορίες των δικαιούχων να προβλέπονται τέτοιοι έλεγχοι. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα απλούστευσης. Εισφορές σε είδος. Αυτού του είδους οι εισφορές θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες και ακόμα και αν δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες, εμείς καλούμεθα να κάνουμε ελέγχου για αυτές τις εισφορές. Απλουστεύουμε και εδώ πέρα την κατάσταση. Αν δεν είναι επιλέξιμες, δεν θα γίνονται εκ των προτέρων έλεγχοι για τις φορές αυτές. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε εδώ πέρα μια άμεση απλούστευση των πραγμάτων. Στο παρελθόν όλες οι οντότητες έπρεπε να υποβάλουν πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Δεν προβλέπεται η απέτηση αυτή όταν δεν προβλέπονται πλέον συγκεκριμένοι κανόνε ή απαιτήσει για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία άμεσα λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση. Να σα δώσουμε και κάποια απτά παραδείγματα όσον αφορά την κατάργηση αυτή των ελέγχων όσον αφορά τις εισφορές σε είδος. Αυτά όσον αφορά τις απλουστεύσεις στη φάση εφαρμογής, στη φάση εκτέλεσης ισχύουν και για το γενικότερο πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου είπαμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε περισσότερο προς ένα ηλεκτρονικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα μας οδηγήσει τελικά και στο σύστημα αυτό των ηλεκτρονικών επιδοτήσεων, όπου θα έχουμε ένα εταιρικό ηλεκτρονικό σύστημα για τους ετούντες, προκειμένου να μπορούν να καταβάλουν τις, να υποβάλουν μάλλον τις αιτήσεις χρηματοδότησης. Και θέλουμε για τη νέα γενιά επενδυτικών προγραμμάτων να έχουμε εναρμόνιση των διαδικασιών και των κανόνων. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται στο πλαίσιο της εναρμόνισης που προβλέπεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ας περάσουμε τώρα στην ε, φάση της πληρωμής, αφού αφήσαμε τη φάση της υποβολής ουσιαστικά της αίτησης. Εδώ πέρα έχουμε μία σειρά από δαπάνε που μπορεί να είναι φάπαξ ποσά, κόστο μονάδο ή αποκοπήν ποσά. Για ποιο λόγο θεωρούμε εμεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εδώ πέρα πιο απλουστευμένε ε, επιλογέ δαπανών. Το κάνουμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερο στα αποτελέσματα, έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνεται επίση το διοικητικό άγχο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάζει κατά αυτόν τον τρόπο μια γενικότερη προσέγγιση που είχε όσον αφορά τι δαπάνε αυτέ. Λέμε πιο συγκεκριμένα ότι ε, είτε μπορούμε τελικά να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα και απλουστεύονται τότε τα πράγματα, ή αν δεν, μπορεί, ο, αν δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε τελικά στα αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχει και μια αιτιολόγηση γι' αυτό. Ποιε είναι τώρα οι πλουστεύσει αυτέ οι οποίε προβλέπονται με μεγαλύτερε λεπτομέρειε, θα τι δούμε. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στι εισρωέ κυρίω. Βλέπουμε ποια είναι τα στοιχεία του κόστου μια δράση. Για παράδειγμα, θα δούμε το κόστο αναμονάδα που καλύπτει δαπάνε προσωπικού για ένα άτομο το οποίο εκπαιδεύει νέου επιχειρηματίε. Στο μέλλον αυτό που μα ενδιαφέρει είναι περισσότερο το αποτέλεσμα. Στα πλαίσια δηλαδή τη εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών, αυτό που μα ενδιαφέρει είναι τα, τα καταποκοπήν ποσά να συνδεδοθούν με το σύνολο του κόστους της κατάρτισης και με το σύνολο των δικαιούχων της κατάρτισης αυτής. Δεν κοιτάμε λοιπόν πλέον τόσο πολύ τις εισρωές όσο τα αποτελέσματα και έχουμε ένα συνολικό καταποκοπήν ποσό που έχει να κάνει με το σύνολο της δράσης αυτής. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα απλούστευσης. Επί του παρόντος είναι το σύνολο των επιτρόπων, το σώμα των επιτρόπων, το οποίο αδειοδοτεί. Στο, μέσο, στο μέλλον θα έχουμε αδειοδότηση από εξοδοτημένο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα περνάμε από δίμηνη περίοδο αδειοδότηση σε μία περίοδο μόνο δύο εβδομάδων. Απλουστεύσει επίση, κληθήκαμε να κάνουμε σε τομεί ε, χρηματοδότηση όπου δεν είχαμε στατιστικά ή ιστορικά δεδομένα. Στο μέλλον κάθε φορά που δεν έχουμε τέτοια δεδομένα θα χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο ονομάζουμε την κρίση, την άποψη του εμπειρογνώμονα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τις απλουστευμένες αυτές μορφές παρουσίας των δαπανών ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές που δεν έχουμε δηλαδή στατιστικά ιστορικά δεδομένα. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το πεδίο εφαρμογή των νέων αυτών απλουστευμένων επιλογών για τι δαπάνε. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένα προγράμματα. Εμεί στο μέλλον λέμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σύνολα δράσεων στο σύνολο των προγραμμάτων και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ θετικό για τους ίδιους τους δικαιούχους. Για παράδειγμα, σήμερα μπορεί να έχουμε μονάδες κόστους για τις ταξιδιωτικέ δαπάνες ανά πρόγραμμα, ενώ στο μέλλον προτείνουμε όλες οι μονάδες κόστους για ταξιδιωτικές δαπάνες να εφαρμόζονται για όλα τα προγράμματα, τα κοινοτικά, στα οποία προβλέπονται δαπάνες ταξιδίου. Με ένα λαπτό παράδειγμα απλούστευσης της ε, ακολουθητές διαδικασίας, η οποία θα επωφελήσει τους ίδιους τους δικαιούχους. Ας δούμε κάποιες άλλες μορφές ε, εισφορών. Έχουμε νέες απλουστευμένες εισφορές, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε τρόπους ε, αποζημίωσης που δεν βασίζονται στο κόστος, αλλά στα αποτελέσματα. Επομένως, η πληρωμή έχει να κάνει με συγκεκριμένη παράδοση αποτελέσματος. Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Ουσιαστικά έχει να κάνει με συγκεκριμένε δράσεις μόνο. Να σας δώσω δύο παραδείγματα προκειμένου. Έχουμε για παράδειγμα δράσεις οι οποίες δημιουργούν κίνητρα αντί ουσιαστικά απλώ να αποζημιώνουν τους δικαιούχους. Για παράδειγμα, δεν θα δώσουμε απλώς μια επιδότηση σε έναν παραγωγό προκειμένου να παράγει κρασί, αλλά θα μπορέσουμε να συνδέσουμε την επιδότηση αυτή με την παραγωγή κρασιού κατά τρόπο αηφόρο, ανανεώσιμο. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε δύο πολιτικές οι οποίες εδώ πέρα επιτυγχάνονται. Και παραγωγή κρασιού, αλλά και καλύτερη χρησιμοποίηση της ενέργειας, για παράδειγμα. Να σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα πληρωμών που δεν έχει να κάνει με τις εισρωές μόνο. Πληρωμές που έχουν να κάνουν με τι συνθήκε που θέτει ο ίδιο ο νομοθέτης για συγκεκριμένε πολιτικές. Για παράδειγμα, στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου μετανάστευση και ένταξη, κάνουμε πληρωμέ ανά πρόσφυγα που έχει μετεγκατασταθεί, χωρί αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να υπολογίσουμε το ακριβέ ποσό υποστήριξη πλαισίωση του πρόσφυγα αυτού. Προβλέπεται ένα συγκεκριμένο καταποκοπήν ποσό στην ίδια την νομοθεσία δηλαδή. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, το οποίο μπορεί να έχει περισσότερο συμβολικό τελικά χαρακτήρα, είναι η ίδια η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλουμε να εμπλακούν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτε στην εκτέλεση του κοινοτικού προπολογισμού σε όλα τα επίπεδα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την ίδια τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, όσον αφορά την κατασκευή συγκεκριμένων υποδομών. Θέλουν τη δημιουργία κάποιου παιδικού σταθμού, θέλουν να δημιουργηθούν κάποια άλλα έργα. Όλα αυτά θα τα λαμβάνουμε πλέον υπόψη μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον πολίτη, ιδίω όσον αφορά την εθελούσα εργασία. Ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μη κυβερνητικέ οργανώσει μα λένε ότι δεν καταμετράται σωστά η εθελοντική εργασία. Εμεί αποφασίσαμε να αλλάξουμε την κατάσταση και να καταγράφουμε πλέον εθελοντική εργασία κατά τον ακόλουθο τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να φέρουμε σε δύσκολη θέση, να ζημιώνουμε τελικά μια μη κυβερνητική οργάνωση επειδή χρησιμοποιεί εθελούσια εργασία. Αντίθετα προσπαθούμε να δώσουμε κάποια κίνητρα και να σας δώσω εδώ πέρα κάποια παραδείγματα. Ας πάρουμε μία, μία κυβερνητική οργάνωση η οποία ασχολείται με δράσεις κατά της διακριτικής μεταχείρισης. Έχουμε το κόστος της δράσης, ας πούμε ότι είναι 100, από τα 100 τα 50 καλύπτονται από τους εθελοντές και έχουμε 30 ευρώ όσον αφορά το προσωπικό και 20 όσον αφορά τις υποδομές. Το συνολικό ποσό είναι 80 και η χρηματοδότηση έφτανε μόνο τα 40 ευρώ. Εμεί προτείνουμε η χρηματοδότηση να φτάσει μέχρι το 80, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν πληρώσει μόνο 50 ευρώ θα φτάνει μέχρι εκεί η χρηματοδότηση. Ουσιαστικά θα καλύπτουμε πλέον τις πραγματικές δαπάνες στις οποίες έχει προχωρήσει ο δικαιούχος, εν προκειμένου μη κυβερνητική οργάνωση. Άρα κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτουν όλες τις πραγματικές τους δαπάνες ως μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά δεν πληρώνουν, αν θέλετε, την λεγόμενη δωρεάν ή μη ε, μισθωτή εργασία και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο εύκολα εθελοντές. Και οι ίδιοι οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών τάχθηκε υπέρ αυτού. Τώρα, η κατάργηση της αρχής της μη δημιουργίας κέρδους. Το ζήτημα αυτό είχε προκαλέσει πάρα πολλά ερωτήματα στο παρελθόν. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια όσον αφορά στην αρχή αυτή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εμεί να καταβάλουμε ποσά την οποία υπερβαίνουν το επιλέξιμο κόστο. Αυτό είναι σαφέ και δεν τροποποιείται. Και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση την συσσόρευση κοινοτική χρηματοδότηση για συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εμεί θεωρούμε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε σημαντικό πρόβλημα γιατί εν προκειμένου τα projects αυτά τα οποία δημιουργούν έσοδα δεν χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένε επιδοτήσει αυτή τη στιγμή, αλλά χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα κινούμεθα ουσιαστικά περισσότερο αυτή τη στιγμή σε χρηματοδοτήσεις όπου δεν υπάρχει δημιουργία κέρδους και όπου ο μόνος τρόπος υποστήριξης τελικά ενός έργου είναι η ίδια επιδότηση. Σε όλε τι άλλε περιπτώσει, όπω σα είπα, υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα. Αναφέρουμε στα προγράμματα εκείνα τα οποία από μόνα τους αυτή τη στιγμή αρχίσουν να εφαρμόζονται, μπορούν να δημιουργήσουν κέρδος. Όπως σα είπα, είχαν προκύψει διάφορα ερωτήματα όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Βλέπετε πόσα πράγματα πρέπει να κάνουμε σήμερα προκειμένου να δούμε ποια είναι τα έργα εκείνα τα οποία δεν μπορούν να δημιουργήσουν από μόνα τους ε, έσοδα. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε το αρχικό κόστος, να δούμε τα συγκεκριμένα τιμολόγια, να δούμε αν υπάρχει κάποιο πλεόνασμα όσον αφορά το επιλέξιμο κόστος, να δούμε τα καταναλογή ε, κέρδη τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν και καταλήγουμε σε ένα τελικό ποσό. Η όλη διαδικασία όμως είναι πάρα πολύ πολύπλοκη Γι' αυτό το λόγο στο μέλλον σας προτείνουμε να διαγράψουμε όλα αυτά τα στάδια τα οποία βλέπετε στη διαφάνεια από το 4 ως το 7. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στις δαπάνες. Βλέπετε εδώ πέρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στην διαφάνεια αυτή. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε ένα ποσό το οποίο υπερβαίνει το αρχικά εγκεκριμένο ποσό της κοινοτική χρηματοδότησης και από την άλλη προσπαθούμε να προστέψουμε την όλη διαδικασία δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα σύστημα το οποίο δεν θα επιβαρύνει ούτε τον κοινοτικό προπολογισμό, αλλά δεν θα δημιουργεί διοικητικό άχθος και για τον ίδιο τον αποδέκτη, τον δικαιούχο. Ένα άλλο σημαντικό τμήμα της πρότασής μας, το οποίο λειτουργεί υπέρ των δικαιούχων, είναι η αρχή της, του ενιαίου ελέγχου. Και πάλι εδώ πέρα θα μπορούμε να έχουμε ελέγχους και από εξωτερικές αρχές και θα μπορούμε να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα υποβολής στη συνέχεια ελεκτικών εκθέσεων. Ξέρετε ότι Μπορεί να έχετε πάει σε τρίτες χώρες όπου οι μη κυβερνητικέ εργανώσεις πάρα πολλές φορές ε, ε, λένε ότι ε, το διοικητικό άκθος το οποίο τους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αυτή τη στιγμή με το ενίο αυτό σύστημα ελέγχου και με τις ενιαίες μεθόδους ελέγχου τα πράγματα πλουστεύονται και μειώνεται πάρα πολύ το διοικητικό άχθος. Και ξέρετε ότι εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις γενικές συμφωνίες που έχουμε με α, σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς ή εταίρους. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε κοινοτικά κονδύλια τα οποία περνάνε σε ένα διεθνή οργανισμό προκειμένου να τύχουν από εκεί πέρα διαχείρισης και να περάσουν σε συγκεκριμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, προβλέπεται εδώ πέρα μια σειρά ελέγχων και παληθεύσεων για την ίδια όμως δράση και για το ίδιο πρόγραμμα. Έχουμε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγχο από το διεθνή οργανισμό, έλεγχο από εσωτερικό ελεκτή, έλεγχο από εξωτερικό ελεκτή, και έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και δεν είναι θεωρητική, θεωρητικό το παράδειγμα αυτό. Για συγκεκριμένα προγράμματα είχαμε δύο και πέντε αλλεπάλληλου ελέγχου. Εμεί αυτό το οποίο σα προτείνουμε είναι να αρχίσουμε να ε, περιοριζόμαστε απλώς στον έλεγχο που κάνει ο τρίτος διεθνής οργανισμός. Ξέρουμε ότι είναι έμπιστος ο οργανισμός αυτός, ξέρουμε ότι ακολουθεί συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα ελέγχου, επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χρήση των κονδυλίων ή του έλεγχος των κονδυλίων θα γίνει σωστά. Αν υπάρχουν βέβαια υποψίες για παρατυπίες στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων, εμείς προφανώς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθουμε και θα κάνουμε τον επιπλέον έλεγχο. Δεν εγκαταλείπουμε αν θέλετε τη δυνατότητα ελέγχου που μας δίδεται. Απλώς δεν υπάρχει λόγο να γίνονται επιπλέον έλεγχοι στι περιπτώσει εκείνες που δεν έχουν εντοπιστεί σφάλματα. Θα ολοκληρώσω στο σημείο αυτό το πρώτο τμήμα τουλάχιστον τη παρουσίασή. μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τόσο ξεκάθαρη παρουσίαση. Πράγματι. Αν εγκρίνουμε προτάσεις τροποποίησης θα υπάρξει λιγότερη γραφειοκρατία. Πρώτα κύριε Γκρέσλερ, η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι εδώ είναι τεράστια δουλειά που μας έχετε παρουσιάσει. Έχουμε πολύ περίπλοκες αλλαγές εδώ στον προϋπολογισμό ως μόνιμη. Η συγκεκριμένη είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσες αλλαγές από το 2005. Μια μεγάλη αλλαγή λοιπόν στα κείμενα που όμως δεν μας αφήνεται αρκετός χρόνος για την επεξεργαστούμε, πράγμα το οποίο δεν το δέχομαι. Πρέπει λοιπόν να τραβήξουμε το φρένο, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες. Έχουμε να κάνουμε με 780, 780 σελίδες πρόταση. Όλα μου τα Χριστούγεννα και τις μέρες της πρωτοχρονιάς με αυτές ασχολήθηκα. Και ε, αισθάνομαι ιδιαίτερη δυσφορία γιατί θα έπρεπε αυτή, ε, αυτό το κείμενο να ε, απλουστεύει συγχωνεύοντας κανόνες δημοσιονομικούς και όρους εφαρμογής που είναι οι λεπτομερείς αυτές οδηγίες προς το προσωπικό προβαίνει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, δηλαδή είναι ερμηνευτικές οδηγίες ουσιαστικά για να γίνεται ομοιόμορφη η ερμηνεία. Τώρα βλέπουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί αυτοί οι κανόνε εφαρμογή, τα rules of application, ώστε να γίνει πιο απλή διαδικασία. Αντιθέτω, έχουν μείνει κάπου εδώ και κάπου εκεί. Ε, έχουν εχωθεί σε κάποια άλλη παράγραφο έχουν ε, ε, εν πάση περιπτώσει συγχωνευτεί και ταυτόχρονα αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία και τελικά δεν είναι τελείως διαφορετική εικόνα του προπολογισμού. Η βασική ε, αλλαγή λοιπόν δεν είναι ότι έχουμε τα παλιά κείμενα. Όχι, έχουμε τα παλιά κείμενα με νέα διατύπωση και διάρθρωση. Έχουμε παραδείγματι τη γενική άδεια για τις χορηγίες από επιχειρήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε, δεν μπορούμε να το εισαγάγουμε έτσι. Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι εύκολο να ανοιχνευτεί πού βρίσκεται το κείμενο, σε ποια θέση έχει πάει το μέχρι τώρα ισχύον κείμενο και χωρίς καμία, καμία εξήγηση για τη μετακίνηση του συγκεκριμένου σημείου, του συγκεκριμένου κειμένου ή κάποια, κάποιο άλλο βάσιμο λόγο. Επομένω είναι πολύ ασαφής αυτή η εικόνα που έχουμε και εγώ έχω δεσμευθεί και έχω προσυλλοθεί στον αγώνα για ένα single rulebook, για ένα και μόνο ενιαίο κανόνα, ένα ε, εγχειρίδιο κανόνων καλύτερα. Ε, δεν το καταφέραμε όμως. Δυστυχώς και με μεγάλη μου δυσφορία διαπιστώνω ότι κάποιοι κανόνες εφαρμογής εξαφανίζονται και καλύπτονται από κατευθυντήριες γραμμές, guidelines, που όμως δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί, δεν έχουν ακόμη διατυπωθεί, μας τις έχουν υποσχεθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν τις έχουμε δει. Και πάλι εδώ θα διαφωνήσω. Και μην ξεχνάμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμέ οι guidelines, δεν έχουν νομική ισχύ, δεν είναι δεσμευτικέ. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα ισχύσουν όχι μόνο στην εκτέλεση του προπολογισμού από την Κομισιόν, αλλά και από όλε τι υπηρεσίε. Επομένω, δεν μπορούμε εμεί να επαφεθούμε στο ότι ο καθένα θα γράφει ότι του έρχεται και θα προβαίνει στην εκτέλεση του προπολογισμού όπω να είναι. Πρέπει να είναι σαφεί η όροι και οι οδηγίες για το πώς διαχειρίζεται ποιος, ποιο κονδύλιο και με ποιο τρόπο. Αυτή είναι η βασική μου επίκριση λοιπόν, ξεκινάω, ότι είναι πολύ ασαφής η εικόνα. Έχουμε τους τομεακούς επίσης ε, κανονισμούς, όπου πάλι δεν κατέστη δυνατόν να ενσωματωθούν στον γενικό κανονισμό. Μας ανησυχούν πολύ όλα αυτά λοιπόν ε, και θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία να έχει δοθεί περισσότερος χρόνος, να γίνει με πολύ μεγαλύτερη προσοχή η προετοιμασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και κάποια χρόνια πίσω μας ήδη. Καταλαβαίνω ποια είναι τα όρια των δυνατοτήτων της Επιτροπής, αλλά πρέπει και εσείς να τηρήσετε κάποια όρια ποιότητα στη δουλειά. Οι ορισμοί, οι ορισμοί είναι μεταξύ τους πολλές φορές αντιφατικοί. Είναι αντιφατικοί ε, είναι αντιφατικός ένα ορισμό με ένα άλλο κείμενο της Επιτροπής. Ε, η μόχλευση, ο πολλαπλασιαστικό παράγων, η αξιοπιστία, η παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, όλα αυτά είναι σαφείς, ασαφείς έννοιες. Και επίσης η προσπάθεια που θέλουμε τελικά να υλοποιήσουμε, δηλαδή προϋπολογισμός για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Budget for results δεν τηρείται ως προσέγγιση, ως προσανατολισμός πάγιος, εμφανίζεται σε κάποια σημεία κάπου χάνεται, κάπου τη λησμονούμε την προσέγγιση αυτή. Λοιπόν, αυτή, αυτός ο προσανατολισμός, η προσέγγιση στο αποτέλεσμα πρέπει καταρχάς να είναι σαφής ως έννοια, τι είναι, πώς προσμετράτε και στη συνέχεια με τρόπο σταθερό και πάγιο να επιδιώκεται μέσα από τα κείμενα. Εγώ θα καταθέσω βέβαια τις σχετικές τροπολογίες για τα δικαιώματα και τις προνομίες του Κοινοβουλίου, πάρα πολύ σημαντικό, στις μεταφορές, τα over. Βεβαίω ε, κατάφερε η Επιτροπή να εισαγάγει περισσότερε εξουσίε για τον εαυτό τη και ε, προσπαθεί να βγάλει κάποιες από τις δικές μας αρμοδιότητες ε, διακριτικά. Σε ορισμένα σημεία δεν θα διαφωνήσω 100% αλλά θα επισημάνω το εξή ότι υπάρχει δυνατότητα στην πολιτική για τα κτίρια κονδύλια εν όλο που προβλέπονται ως δαπάνες για ε, την κτηριακή πολιτική και τα κτίρια να μπορούν να μεταφερθούν. Έχουμε πει όμως ότι δεν είναι δυνατόν να πληγούν οι αρχές, οι βασικές αρχές της δημοσιονομικής πολιτικής που χαρακτηρίζουν τον προπολογισμό. Το ενιάφσιο, παραδείγμα του προπολογισμού, δεν μπορεί μέσω αυτής της επιλογής για μεταφορά κονδυλίων να ε, πληγεί. Καταπιστεύματα. Καταρχάς πρέπει να διερωτηθούμε, τα θέλουμε, γιατί εκεί δεν μπορούμε να ελέγξουμε καθόλου την ε, εφαρμογή τους και την εκτέλεσή τους. Καλή άλλωστε εμπειρία από τον έλεγχο του προϋπολογισμού δεν έχουμε εν προκειμένου. Και άρα θέλουμε πιο πολλές πληροφορίες ε, για το, και από εσά για το πώς θα σταθούμε στην υπόθεση αυτή και αυτό βεβαίως όπως είπα πλήττει και βασική αρχή του προϋπολογισμού εν προκειμένου του ενιαίου προϋπολογισμού. στις ε, δωρεές, οι χαριστικές αιτίες, όπου είναι η Ένωση ε, ο κύριος χορηγός, μπορούμε να έχουμε πιο ελαστικούς κανόνες σε σχέση με τον έλεγχο, αλλά πρέπει να τηρούνται απαρέγκλητα οι υποχρεώσεις λογοδοτησίας για τους λοιπούς οργανισμούς και φορεί. Δεν πρόκειται να δεχθούμε γουρούνι στο σακί. Για τους λοιπούς φορείς θέλουμε ξεκάθαρους κανόνες και λογοδοσία. Χορηγίες από εταιρείε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το ξαναδούμε αυτό. Ένα σημείο όμως που θέλω να αναφέρω είναι το σχετικό με την ε, εισαγωγή ανάλογα και με το επίπεδο της ε, διαχείρισης μιας εξωτερήκευσης των πόρων, δηλαδή θα προέρχονται από εξωτερικούς φορείς, την οποία δεν έχουμε προβλέψει και δεν θέλουμε. Επομένως, τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή, θα έχει το ρόλο ενός διοικητικού συμβουλίου. Ποιος θα ελέγχει. έμεση διαχείριση, service level agreements. Εδώ θα ήθελα να ξέρω τι εννοεί η Επιτροπή με την πρόταση για συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιακό. Δηλαδή, γενικέ διευθύνσει θα έρχονται απευθεία σε συνεννόηση κάθε μία με έναν εξωτερικό παράγοντα, μια υπηρεσία αποκεντρωμένη ή ακόμη και άλλου φορεί και δεν θα υπάρχει καμία παρέμβαση της Επιτροπής ως συλλογικού οργάνου, δηλαδή θα είναι σε επίπεδο ισότιμο γενική διεύθυνση με εξωτερικό παράγοντα ε, και θα λαμβάνει έτσι τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και την εκτέλεσή του. Νομίζω ότι είναι τόσο σαφείς οι διατυπώσεις που αφήνουν μεγάλο περιθώριο στη φαντασία. Και θα θέλαμε να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στις ε, ε, προμήθειες. Εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να δω η εσωτερική αγορά τη γνώμη έχει, γιατί πιστεύω ότι έχει τη σχετική ε, πραγματογνωμοσύνη και θα μπορούσε να μας στηρίξει. Αλλά δυστυχώς δεν θέλησαν να μας κάνουν καμία έκθεση και έτσι θα στερηθούμε τις πολύτιμες συμβουλές τους. Πάντως υπάρχουν ε, πολλά θέματα που μπορούν οι συνάδελφοι να μας ε, δώσουν ως πληροφορίες. Και βλέπω ότι πολλά πάνε στα παραρτήματα εδώ. Επιλογές κόστους στην πρόταση. Απλουστευμένες επιλογές κόστους σημαίνει ότι θα πάντοτε από τον δικαιούχο που πάντα θα έχει καλύτερες εκδοχές αποδείξεως του κόστου σε σχέση με το πραγματικό. Αντιφάσεις επίσης βλέπω σε σχέση με ε, διάφορα σημεία του κειμένου. Άλλος είναι ο εντολέας, δηλαδή, της ε, δαπάνης και άλλος είναι ο υπεύθυνος προς εκτέλεση αλλά ταυτόχρονα μας λέτε ότι θέλετε να ε, καταστήσετε πιο απλές τις συνθήκες για τους δικαιούχους. Εδώ βέβαια καταλαβαίνω ότι υπάρχει προσπάθεια να καταστεί πιο εύκολο το έργο του εντολέα και ο κάθε εντολέας ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ε, ο authorizing officer, ότι θα προσπαθεί πάντοτε να καλύπτεται στο δυνατόν περισσότερο, αλλά δεν είναι δυνατόν και να εκμηδενιστούν τα πάντα. Δεν σκοπεύω μάλιστα να κάνω πάρα πολλέ ε, τροπολογίε, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ να το κρύψω, θα υπάρξουν κάμποσε. Εγώ με πάντοτε υπέρ τη απλούστευση. Αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν το ιστορικό τους, το λόγο για τον οποίο έχουν μπει στο κείμενο, μπει στα προηγούμενα κείμενα. Και ξαφνικά βλέπουμε με μια μονοκοντιλιά να διαγράφονται. Αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε ότι υπάρχουν άρθρα τα οποία έχουμε συζητήσει επί ώρες. επί ώρες για να συζητηθούν και να ενταχθούν στα κείμενα και μετά χωρίς κανένα περιθώριο για συζήτηση, χρονικό ή μη τι άλλο, βλέπουμε να διαγράφονται. Ε, αυτά όλα θα τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Πρέπει βεβαίως να ε, δούμε τις θέσεις και της Επιτροπής των Προϋπολογισμών. Η δική μου θέση και εντύπωση είναι μεικτή θα έλεγα. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα έναντι αντιδράσει καλύτερα έναντι των προτάσεων αυτών σε άλλα σημεία θα μπορούσα να το δεχθώ, σε άλλα νομίζω όχι και εν πάση περιπτώσει χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να τα μελετήσουμε. Ευχαριστούμε. Κυρία Κρέσελ, προφανώς περάσατε τις διακοπές διαβάζοντας. Ευχαριστούμε πάντως. Έτσι επιστρέφουμε στην πραγματικότητα. Μπράβο, η πραγματογνωμοσύνη σας μας είναι πολύτιμη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριο Σάσουαρθ να σχολιάσω κάποια ζητήματα που τίθενται στο πρώτο μέρος της έκθεσης αυτής, αλλά προηγουμένως θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, για το θέμα της απλοποίησης συνολικά. Φυσικά και το καλοδέχομαι και τα σχόλια της κυρίας Γκλέσσερ. Εγώ ήμουν εισηγητή στην προηγούμενη εντολή για την απλοποίηση όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Έχω πιστεί ότι η απλοποίηση είναι απολύτως αναγκαία για τους δικαιούχους, ότι έχουν πιο εύκολο και πιο γρήγορα πρόσβαση στα κονδύλια, ότι είναι κάτι ουσιαστικό επίσης και για την διοίκηση, αλλά και πιο συγκεκριμένα έχει αποδείξει ότι μειώνει και το περιθώριο σφάλματος. Και αυτό είναι στόχος μας. Οπότε Θαυμάζω τα σχόλια σχετικά με την αλλαγή νοοτροπίας που συνάδουν απόλυτα με την απλοποίηση. Ένα δεύτερο σχόλιο όμως που έχω να κάνω από την άλλη έχει να κάνει με τις πολιτικές μας των προηγούμενων ετών. Και γιατί η πολιτική μας όσον αφορά την επίδοση του προπολογισμού. Εντάξει, λέμε ότι θα μας βοηθήσει να χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους, αλλά πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι δείκτες επιδόσεων. Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνουν αυτοί οι δείκτες. από τη μια και από την άλλη, η ανησυχία είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα σε αυτούς τους δείκτες επιδόσεων και την απλοποίηση γενικότερα του προπολογισμού. Πρέπει να το συζητήσουμε πολύ περισσότερο για να είμαστε σίγουροι για το τι θέλουμε να πετύχουμε όταν μιλάμε για προπολογισμό βασισμένο σε επιδόσεις. Και συγχρόνως θέλουμε και απλοποίηση. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν στηρίζω το ένα ή το άλλο. Τα στηρίζω και τα δύο. Απλώς μην υποτιμάμε τη δυσκολία που θα συναντήσουμε προκειμένου να τα πετύχουμε αυτά. Η κυρία Κρέσλερ Όντω, μα εξήγησε την πολυπλοκότητα. Εγώ δεν πέρασα τα Χριστούγεννα μελετώντα αυτό το θέμα, πρέπει να το ομολογήσω. Είναι όντω περίπλοκο. Και εδώ μπαίνουν μαζί τόσε διαφορετικές επιτροπές, αυτό είναι απόδειξη. Και άντε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα έγκαιρα. Τώρα όσον αφορά την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία, ευχαριστώ τους συναδέρφους Κάτι που βγαίνει από το πρώτο αυτό τμήμα. Η αρχή μη κέρδους και θα ήθελα να εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λογική πίσω από αυτό. Χρειαζόμαστε να μας καθισχάσει περισσότερο. Για το πρόγραμμα ενιαίου ελέγχου. Εγύρει ζητήματα. Ποιος ελέγχει κατά πόσο υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον κανονισμό. Payment Bond Delivery. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει να αναγνωρίσουμε ότι έχει περιορισμένες, ε, περιορισμένα αποτελέσματα. Και επίσης η μικρότερη χρονική διάρκεια. Η έκθεση μιλάει για την κρίση εμπειρογνωμόνων. Ναι, αλλά ποιο είναι εμπειρογνώμων για να κρίνει. Και τέλος, από αυτό το πρώτο τμήμα, στη δεύτερη διαφάνειά σας, αναφέρεστε σε φυσικά πρόσωπα. Και τι είναι ένα μη φυσικό πρόσωπο. Αυτά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σουλίνη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα επιτρέψει περισσότερη ευελιξία στην διαχείριση του προπολογισμού και απλοποίηση για τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είχε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Όταν επιβεβαιώσαμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από τέσσερα χρόνια, δεν υπήρχε πρόβλημα με την μετανάστευση κτλ. Είχαμε, είχαμε τότε μόνο το 3% των ε, κατοίκων που ήταν ε, μετανάστες. Τώρα όμως γίνονται σοβαρά ζητήματα για τους πολίτες όσον αφορά την ανεργία. Το 45% των πολιτών θεωρούν ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετανάστευση δηλαδή. Και σε δεύτερη θέση έρχεται η τρομοκρατία με 30% των Ευρωπαίων σύμφωνα με το βαρόμετρο να θεωρούν ότι είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Συνεπώς πρέπει να δράσουμε γρήγορα για να ανακτηθεί και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι ξέρουμε ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη, κάτι το οποίο είναι προς όφελος των λαϊκιστών και μόνο. Στην ε, Σλοβενία λέμε ότι αυτός που δίνει γρήγορα δίνει δύο φορές. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας στον προπολογισμό. Χρειάζεται απλοποίηση των κανόνων για την χορήγηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και χαίρομαι που έχουμε αυτή την πρόταση. Όταν βρίσκομαι με τους εκλογείς μου, τους ψηφοφόρους μου, με ρωτούν συνέχεια ποιες είναι οι διαδικασίες, γιατί είναι τόσο περίπλοκες. Κάποιοι, μάλιστα, έχουν και κάποιες θεωρίες συνωμοσία. Λένε ότι οι διαδικασίες επίτηδες είναι τόσο περίπλοκες, ώστε οι πολίτες να μην μπορούν να δικαιούνται κονδύλια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να τους δίνει. Συνεπώς, η απλοποίηση είναι σημαντική και όλοι συμφωνούμε από αυτού. Αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί όταν προχωράμε σε απλοποίηση. Να υπάρχει διαφάνεια και να είμαστε και αποτελεσματικοί, κάτι το οποίο είπαν ε, και οι συγητές. Πέρυσι επετέχθη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ότι η νομοθεσία θα πρέπει να είναι καλύτερη νομοθεσία. Πράγματι, δεν θέλουμε παραπάνω διοικητικό άχθος. Θέλουμε η νομοθεσία μας να είναι πρακτική και να εφαρμόζεται εύκολα. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή αποτελεί ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί μιλάμε για απλοποίηση και εναρμόνιση. Όμως μας μένει πολλή δουλειά ακόμα, αν θέλουμε να έχουμε μια διαχείριση βασισμένη σε επιδόσεις. Έρχομαι τώρα στους ενιαίους ελέγχους και πώς μπορούμε να βασιστούμε στον έλεγχο άλλων ε, οργάνων. Πώς θα είμαστε σίγουροι ότι οι έλεγχοι των διεθνών οργανισμών είναι υψηλών προδιαγραφών και κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Σαρβαμά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, φιλόδοξη πρόταση που μας έκανε. Θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια την κυρία Γκρέσλε για το ότι ό,τι και αν κάνουμε όσον αφορά τα αποτελέσματα βάση επιδόσεων πρέπει να πηγαίνουμε στο βάθος του προβλήματος. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Πρέπει να φτάνουμε στο κόκαλο. Το έχω ξαναπεί ότι αυτό το εγχείρημα θα μπερδέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατανόηση αν μόνο επιφανειακά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτήν την τόσο φιλόδοξη ιδέα του να βασιζόμαστε σε επιδόσεις. Αυτό είναι ένα. Και υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να υπενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ το σώμα το 2015 με μεγάλη πλειοψηφία σε μια ολομέλεια ευλόγησε την έννοια της επέκτασης της βάση επιδόσεων αυτής της αρχής και στους ελέγχους. να ισχύει η αρχή αυτή του βάση επιδόσεων και στους ελέγχους. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο μερικές φορές. Στη Γεωργία, για παράδειγμα, δεν περιμένω κανέναν να μετρήσει ποσοτικά τα αποτελέσματα τι βάζουν στην αγορά οι Γεωργοί. Αυτό όμως που περιμένω είναι ότι η ιδέα υπέρ της οποίας ήταν μεγάλη πλειοψηφία και που λέει ότι στις χώρες μέλη όπου υπάρχουν συστήματα που σαφώς λειτουργούν, ε, περιμένω λοιπόν και αυτά να ληφθούν υπόψη για να κρίνουμε το πώς ε, εφαρμόζονται οι έλεγχοι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κατά τα άλλα, δύο λόγια μόνο για τους ε, εισηγητές και συνεισηγητές. Όλοι είναι πολύ καλοί τζεντάι. Η δύναμη να είναι μαζί σας. May the force be with you, είπε ο κύριος Σαρβαμά. Ευχαριστώ κύριε Σπυρίνσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος όσο το δυνατόν. και θα αναφερθώ στις κύριες προτεραιότητες. Ένα που ανέφερε η κυρία Γκρέσλε ήδη, ε, επεξεγηματικό μνημόνιο είναι η πηγή. Εκεί που αναφέρεται ότι οι κύριες διατάξεις των κανονών εφαρμογής μετακινούνται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ενώ λιγότερο σημαντικά στοιχεία θα ενσωματώντα του εσωτερικού κανόνε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι κατευθυντήριε γραμμέ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περίπτωση. Διαφωτίστε μας, ποιος θα αποφασίσει τι είναι το κέριο, τι δεν είναι, τι πάει στους εσωτερικούς κανόνες, τι πάει στις κατευθυντήριες ε, ε, οδηγίες, τι είναι η εσωτερική κανόνας; Πείτε μας να καταλάβουμε και εμείς γιατί έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεύτερον, η απαλφή του, της αρχής ε, της μη κερδοσκοπικής, του μη κερδοσκοπικού φορέα. Ήδη βεβαίως έχουν εκφραστεί σχετικές ανησυχίες και επιφυλάξεις. Πάντως στην ε, διαφάνειά σας για την αρχή αυτή έχετε βγάλει το 4 και 5, δηλαδή προσδιορισμό των αποδεικτικών εισπραξής. Μόνο ορισμένα λέει θα είναι αποδεκτά και μάλιστα δεν θα χρειάζεται να προσφέρονται αυτά που έχουν να κάνουν με το κέρδος. Δηλαδή πώς θα βγάλετε την αρχή του κερδοσκοπικού εάν δεν ξέρετε ότι όντως δεν είναι κερδοσκοπικός ο φορέας. Τρία. Αυτό με τους ενιαίους κανόνες που θα διευκολύνουν ε, την συνεργασία μεταξύ καταπιστευμάτων χρηματοοικονομικών μέσων. Στα καταπιστεύματα. συγγνωμιστά δάνεια. Θα είναι συμπληρωματικά προς τα χρηματοοικονομικά μέσα εφόσον εντάσσονται σε μια ενιαία δράση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα πάντως έχουν ήδη μπει σε, μια, σε ένα σύνολο κανονισμών, έχουν τις αρχές τους, τον τρόπο λειτουργία τους και διερωτώ θα, θα είμαστε πιο πολύ στα χρηματοοικονομικά μέσα, πιο πολύ στον ε, δανεισμό. Πώς έχετε κάνει τις επιλογές σας και ποιος σας είπε ότι οι επιλογές σας θα γίνουν δεκτές. Χρηματο... Ε, καταπιστεύματα. Εδώ ανοίγει πεδίων λαμπρών. Εγγραφή σπόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας γεννά πολλά ερωτηματικά και απορίες. Καταρχάς μιλήσατε για μια σαφή εικόνα της ιστορικής και της εξωτερικής δράσης. Μετά μας είπατε ότι μπορούν τα καταπιστεύματα να θεσπιστούν και για ιστορική δράση και μετά πάτε στα παραρτήματα για να πείτε ότι και για την ενέργεια ακόμα. Μια από τις κύριες πολιτικές που επουδενή δεν είναι δυνατόν να μετακυλιστεί στην χρηματοδότηση από καταπίστευμα. Έχει δικούς τους κανόνες, έχει τραπεζικό λογαριασμό υπάρχει επιτήρηση. Και μάλιστα από το Κοινοβούλιο. Δημοσιονομικό έλεγχο. Και επίσης Μυστήριο για μένα αποτελεί η προθέσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικά το τι εννοεί στο τέλος εκεί. Αν μιλάει για υλοποίηση ή για διαχείριση, implementation in management. Ενώ στην αρχή μιλάει για management, στο τέλος την ξεχνάει τη λέξη. Και στον κανονισμό βλέπουμε τον ορισμό διαφόρων τύπων υλοποίησης ή εκτέλεση Ε, με κοινή implementation. Αλλά μετά μιλάτε για κοινή διαχείριση, έμεση διαχείριση, ε, μεικτή διαχείριση. Μετά μιλάτε για έμεση εκτέλεση. Και κάπως φαίνεται σαν να ε, αφήνει, να μπαίνει στο περιθώριο μόνη της η Επιτροπή σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού γιατί αναφέρεται σε φορείς και πρόσωπα που διαχειρίζονται τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή εκτελούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Φαίνεται σαν μόνη της να παρετείται από τις ευθύνες περί εκτέλεσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μιλάει για άμεση ή κοινή διαχείριση κονδυλίων. Και για να ολοκληρώσω. Αυτή η τόσο φιλόδοξη προσπάθεια νομίζω ότι ισοσκελίστε μόνο από τον τεράστιο αριθμό, εξίσου τεράστιο αριθμό, πάρα πολύ ασαφών καταστάσεων και ερωτηματικών που προκύπτουν από αυτές. Ακόμα και σε αυτό που ανέφερε και η τα ποσά είναι τελείως ακατάλληλα. Ο κύριο Σαρβάμα εξέφρασε το φόβο ότι μπορεί να ε, βελτιώνεται η κατάσταση, να οδηγούμαστε σε μια τερατογένεση κύριος Όλμπριχτ τελευταίος. Πρόεδρε, ευχαριστώ ορισμένες ε, παρατηρήσεις. στην αρχή είχε δοθεί εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο περιμένει τη διαπραγμάτευση για τον Brexit και ότι τίποτα δεν γίνεται. Και ξαφνικά χωρί να έχει αρχίσει διαπραγματεύσει για τον Brexit. Που ούτω ή άλλω όμω δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό, γιατί μπορεί να επηρεάσει τελικά τα αποτελέσματα αυτό. Ε, βλέπουμε ξαφνικά να πιέζει ο χρόνο και να πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα πριν το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί αυτό χρειάζεται να έχει μια βάση σταθερή για να προχωρήσει. Και δεύτερον, εάν η Ίγκεμπορκ Γκρέσλε η ίδια δεν μπορεί να παρακολουθήσει, εμείς οι δόλοι τι να πούμε. Τρίτον, νόμιζα ότι φτάνει τα αγγλικά μου. Γιατί δεν καταλάβαινα το κείμενο. Αλλά εδώ έχουμε γλωσσομαθή... Ε, ε, αγγλόφωνους ε, από μητρική γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν το κείμενο, αλλά μάλλον φταίει η ιδιόλεκτος των Βρυξελών που χρησιμοποιήθηκε. Και για να περάσω στα υπόλοιπα. Έχουμε πολλά ζητήματα που έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα. Και μπορούμε να δώσουμε λύσεις πρακτικές, τεχνικές για το πώς μπορούμε να τα διευθετήσουμε. Αφενός. Αφετέρου υπάρχουν θέματα καθαρά πολιτικής βαρύτητας, υψηλής πολιτικής βαρύτητα. και εκεί πρέπει να δούμε ακριβώς τι προθέσει υπάρχουν πίσω από αυτά, Ποιο τα αποφάσισε. Αυτό που αναφέρατε για εκτέλεση και διαχείριση, άμεση, έμεση, μεικτή, ε, καταπιστεύματα, ε, ένα σειρά, μια σειρά από ε, διαφορετικές ε, ε, διαφορετικούς φορείς. Σήμερα, τα απόγευμα, σήμερα τώρα δεν έχουμε αυτό το θέμα για τους γαλαξίες των ταμείων και τα λοιπά, τόσο σε περίπλοκο αυτό το στερέωμα δηλαδή της χρηματοδότησης. Ε, είναι δυνατόν να επιδεινώσουμε ακόμα τα πράγματα. Επίσης, οι δείκτες για την ε, προσθέμενη αξία. Πώ μπαίνουν εδώ μέσα, δεν είναι θέμα των οικονομολόγων, δεν πρέπει ο ένας οικονομολόγος να το κρίνει πρώτα απ' όλα. ή Είναι κάτι το οποίο ο πολιτικό θα αποφασίσει. Και πώ θα πάρει ο πολιτικό αποφάσει με βάση κάποιου δείκτες. Διαρθρωτικά ταμεία. Έναντι του έτσι. Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Μα όποιο έρθει από την Επιτροπή να μα μιλήσει, μα δεν είναι και άλλη εικόνα. Άλλοι μας λένε, μα κοιτάξτε, όχι, κλειδώνουν μεταξύ τους, είναι συμπληρωματικά. Άλλοι, όχι, όχι, όχι, είναι άλλο πράγμα, μην τα κοιτάτε καθόλου μαζί. Είναι χώρια ή δεν είναι, είναι συμπληρωματικά ή δεν είναι. Αυτό είναι ένα απλό τεχνικό πράγμα. Το θέμα δεν είναι αν θα δέσουμε το έτσι πάνω στα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε. Μην σας παραθέσω τα λόγια των εκπρόσωπων τη Επιτροπή. Χθε ακόμα ήμουν στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου μα είπε ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή ότι δεν έχει καμία σχέση πολιτική συνοχή με το ΕΤΣΕ, αλλά βέβαια είναι συμπληρωματικό γιατί μπορούν να μεταφερθούν κονδύλια από τη συνοχή στο ΕΤΣΕ. Ε, βεβαίω, αν κάποιο θέλει μπορεί να τα μεταφέρει. Για πείτε μου σε πολιτικού όρου τι σημαίνει αυτό. Εάν θέλει μπορεί να μεταφέρει κονδύλια. Είναι τεχνικό το ζήτημα, δηλαδή είναι πολιτικό. Και εν κατακλείδη. Θα συμφωνήσω με την Ingeborg είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο οριζική αλλαγή και αυτό μπορεί να αποτελεί πηγή αισιοδοξία. Είναι πραγματική αλλαγή, δεν είναι τα, τα τεχνητά αυτά ε, εξοραϊστικά σημεία που τα φτιάχνανε το κείμενο, τελικά το περιπλέκανε, που έχουμε δει στο παρελθόν. Είναι ουσιαστική αλλαγή, αλλά θέλει πάρα πολύ προσεκτική ανάλυση και πάντως σαφείς πολιτικές επιλογές από το Κοινοβούλιο για το πώς θέλουμε το επόμενο διάστημα να προχωρήσει. Και ξεκάθαρο διαχωρισμό θέλω να αναφέρω. Χρειάζεται οπωσδήποτε τα τεχνικά να διαχωριστούν από τα πολιτικά ζητήματα και ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής Στάραν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω εγώ δεχομένω στον κύριο Όλμπριχτ, ο οποίος είπε πού πάμε με την πρόταση αυτή. Και διαισθάνομαι εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μειώσει τελικά τους ελέγχους και να μειώσει την νομοθετική δύναμη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι θετικό για τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά βέβαια είναι εις βάρος σαφώς της ίδιας της φύσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και προφανώς θα πρέπει εμείς να αντιταχθούμε σε τέτοιες στάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της συγκεκριμένη πρότασης. Κύριο Σαλή το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε σε έναν ωκεανό εγγράφων και πλέουμε. Ευτυχώς που έχει αναλάβει την εισήγηση η κυρία Γκρέσλε που τα ξέρει τα πράγματα. Τώρα πολύ συγκεκριμένα. 350 σελίδες μας δόθηκαν εχθές μόλις προφανώς δεν είναι σοβαρό να περιμένει κανείς να τις έχουμε μελετήσει. Βεβαίως, καλώς ορίζουμε όλοι ε, τη βασική αρχή της ανάγκης απλούστευσης αυτών των διατάξεων. Πολιτικό θέμα. Και βεβαίως η πολιτική πρέπει να εκφράζεται και με πρακτικό τρόπο. Λιγότεροι κανόνες σημαίνουν ταυτόχρονα και λιγότερα ασφάλματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ο καθένας τους κανόνες να τους ερμηνεύει όπως του αρέσει ή τον βολεύει. Στην παρουσίαση που ακούσαμε σήμερα βλέπουμε μία προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σπρώξει τις, αρμο... τις ευθύνες της στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θα ρωτήσω όπως και οι άλλοι, τι σημαίνει ε, μεικτή διαχείριση. Στην τέταρτη διαφάνεια, επί παραδείγματι, ε, εκεί που λέτε ότι τις ευθύνες για την ε, μεικτή διαχείριση την αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Και αν είναι πολύ περιοριστική, πολύ συσταλτική η εθνική νομοθεσία, τι γίνεται. Πώς θα εκτελεστεί το ποσό. Γιατί βέβαια ο τελικό αποδέκτη χρειάζεται τα ποσά και χρειάζεται και τα κράτη-μέλη να, κάνουν, να ε, λάβουν σχετικές αποφάσεις. Είναι δυνατόν όμως να αφήσει την ευθύνη των αποφάσεων αυτών η Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει πρακτική υλοποίηση. Στην ε, δέκατη διαφάνεια της παρουσίασης έχω την εξή απορία. Ποιος θα ακρίνει εάν είναι ε, έμπειρος επαρκή ειδικός ε, ο αρμόδιος για να κάνει τη σχετική αίτηση και να στήσει τη συνενίσχυση κτλ. Δέκατη τρίτη διαφάνεια. Ο πολίτης πώς θα εμπλακεί όλα αυτά. Θα λαμβάνει αποφάσεις, θα έχει μερίδιο της ευθύνης, Συγκεκριμένα τι εννοείται εμπλοκή των πολιτών. Τι είναι αυτές οι διαβουλεύσεις, θα κάνετε δημοψηφίσματα. Βασικά είναι αυτά τα ερωτήματα, αλλά πρέπει να δώσετε Δεκατιένατη 19η διαφάνεια. Καλή σαν ιδέα μεν, ε. αλλά πάλι το ζήτημα αξιοπιστίας. Εδώ μιλάτε για ε, εκτιμήσεις και μετά κρίσεις. Με την ενιαία αυτή ε, λογιστική επαλήθευση, το single audit, θα έχετε και έναν κατάλογο των φορεών εκείνων που θα προβαίνουν στη λογιστική επαλήθευση, στον έλεγχο. Και αν ναι, αυτοί οι φορείς θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες όλοι. Και δει αυτοί οι κανόνες θα είναι εκείνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως είπαν και οι συναδελφοί νωρίτερα, η διαχείριση πώς μεταφέρεται στα κράτη-μέλη, πώς ανατίθεται στα κράτη-μέλη, επί την βάση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν θα είναι απλά τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά τι βλέπουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο μοιράζει χρήματα και που θα ήθελε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί κατά αυτόν τον τρόπο, έχοντας όμως ότι διασφάλιση ότι τηρούνται όλες οι βασικές αρχές ε, της χρηματοδοτικής διαχείρισης με όλους τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Συνεπώς, θέτουμε κανόνες, κανόνες επικανόνων και μετά βέβαια μας προκαλεί εντύπωση ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση ότι αυτοί που ζητάνε ευρωπαϊκά κονδύλια ουσιαστικά γανακτούν και δεν αντέχουν άλλο όλο αυτό το σημαντικό γραφειοκρατικό άχθος που έχει δημιουργηθεί. Νομίζω λοιπόν ότι από την εποχή της Επιτροπής Αντέρ μέχρι σήμερα έχουμε τη συσσόρευση όλων αυτών των διαφορετικών κανόνων που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε προκειμένου να μην μπορούν να μας προσάψουν πλέον τίποτα. Θεωρώ ότι οι ίδιοι υποπέσαμε σε αντιφάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά διορατικοί και κάποια στιγμή να αναλάβουμε και ένα κάποιο ποσοστό ρίσκο αν θέλετε και να έχουμε και μια κάποια εμπιστοσύνη στο σύστημά μας. Διαφορετικά δεν θα βγάλουμε πέρα. Νομίζω πάντως ότι η περιπέτεια αυτή που μας περιμένει είναι καταπληκτική και το εγχείρημα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, η έννοια του φυσικού προσώπου. Κατά την άποψή μου, πως καταλαβαίνω εγώ τον όρο αυτός Γάλλος πολίτης, Ουσιαστικά συνήθω αντιπαραθέτουμε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Νομικό πρόσωπο τι είναι ένας σύλλογο, ένα θεσμός, μια επιχείρηση, μια εταιρεία. Όσον αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία, τα trust funds, έχουμε ένα εργαστήρι σήμερα το απόγευμα. Δημιουργούμε καταπιστευματικά ταμεία, διότι δεν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια μέσα στον προπολογισμό και άρα δημιουργούμε επιπλέον επιπρόσθετα ταμεία αλλά προσέχουμε γιατί πολύ συχνά χάνουμε τελικά τον έλεγχο, ιδίως όσον αφορά τα ταμεία αυτά τα οποία βρίσκονται εκτός κοινοτικού προπολογισμού. Πρέπει λοιπόν κάπου να θέσουμε κάποια όρια. Διαφορετικά δεν θα έχουμε καθόλου τον έλεγχο της κατάστασης. Σε καμία περίπτωση θα ήθελα τώρα να αρχίσω να μιλάω για ζητήματα που θα καλύψουμε σήμερα το απόγευμα. Τούτων λεχθέντων πάντως, νομίζω ότι όσα είπαμε σήμερα το πρωί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, θέλω να ελπίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για Τη Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω το εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρίσκεται εδώ πέρα. Ήρθε με τι καλύτερε δυνατέ προθέσει. Θέλει προφανώ να σημειώσουμε πρόοδο και όπω είπε και η κυρία Γκρέσλε, α μην δημιουργήσουμε ένα νέο πολύπλοκο σύστημα εδώ πέρα. Κύριε εκπρόσωπε λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε να απαντήσετε στι ερωτήσει που ε, τέθησαν από του συναδέλφου και έχουμε να ακούσουμε και το δεύτερο τμήμα τη παρουσίασή σα, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όντως οι παρατηρήσεις ήταν πάρα πολύ καλές και όντως πρέπει να γίνει μια συζήτηση όσον αφορά τη νέα αυτή πρόταση απλούστευσης των δημοσιονομικών κανόνων και απλούστευσης των ελέγχων. Πού θέτουμε τα όρια. Ας μην ξεχνάμε καταρχάς ότι όλοι μας επηρεάζουμε το σύστημα άμεσου ή άμεση ή έμεση διαχείριση, ενώ δεν επηρεάζουμε καθόλου με τι αποφάσει με αυτή τη στιγμή τη λεγόμενη μεικτή διαχείριση. Όπω σα είπα, υπάρχουν κανόνε που θα ισχύουν μόνο για την επόμενη γενιά των προγραμμάτων. Δεν μεταφέρουμε καμία ευθύνη αυτή τη στιγμή προ τα κράτη-μέλη. Όταν αφαιρούμε ένα επίπεδο ελέγχου, ουσιαστικά αφαιρούμε ένα επιπλέον έλεγχο κοινοτικού συγγνώμη, ένα επιπλέον επίπεδο κοινοτικού ελέγχου. Δεν δημιουργούμε νέε ευθύνε ή επιπλέον αρμοδιότητε για τα κράτη-μέλη. Άλλοι μα είπαν ότι σε κάποια άλλα σημεία δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Ας μην ξεχνάμε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο ελέγχων αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή όλους τους κανόνες. Προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε τους περισσότερους κανόνες ως προς τη νέα πρόταση απλούστευσης που έχει γίνει. Όσον αφορά τώρα τις επιχορηγήσεις, δεν προτείνουμε εδώ πέρα κάτι το οποίο είναι ανήκουστο και εξαιρετικό. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τα όσα κάνουν ήδη τα κράτη-μέλη, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε εδώ αναλογικότητα, ισότιμη μεταχείριση, διαφάνεια διαφάνεια, μη διακριτική μεταχείριση, δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και θα πρέπει να καταγράφονται όλοι οι χορηγοί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να βλέπουμε επίσης και όλες τι επιδοτήσεις, όλες οι επιχορηγήσεις, είτε γίνονται ε, σε χρήματα, είτε γίνονται σε είδος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τεθεί ένα νέο πλαίσιο για όλα αυτά. Όσον αφορά τα κτίρια, και εδώ πέρα πάλι δεν κάνουμε σημαντικές τροποποίησεις. Απλώς λέμε είναι πιο εύκολο να δανειοδιοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, αγορά ενός νέου κτηρίου, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κτίρια τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα. Δεν νομίζουμε ότι είναι λογική η πρακτική αυτή από δημοσιονομικής πλευράς. Θα θέλαμε λοιπόν μαζί σας να επανασυζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Και έπειτα ετέθηκε ένα ζήτημα όσον αφορά το σύστημα πώληση κτηρίων, όπου απαιτείται η προαδιοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εσείς ουσιαστικά έχετε κάθε δυνατότητα να κάνετε ελέγχου ή να απορρίψετε την πώληση ενό κτηρίου. Όσον αφορά το single audit, το ενιαίο σύστημα ελέγχων, πάλι εδώ πέρα θα υπάρχει ένα κοινό πυλώνα, που θα συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν όσον αφορά τους ελέγχους. Μόνο εφόσον κληρούνται όλοι αυτοί οι κανόνες θα αρχίσει να εφαρμόζεται και το ενιαίο σύστημα ελέγχου. Δεν θα έρθει το ενιαίο σύστημα ελέγχου να αντικαταστήσει τους ίδιους υφιστάμενους κανόνες. Όσον αφορά το ζήτημα της ε, διαφάνειας, θα δείτε και στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση μείωση των ε, εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται όσον αφορά τη διαφάνεια. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή, χρησιμοποιούμε τον όρο implementation στα αγγλικά γιατί αυτό ακριβώς λέει και η συνθήκη. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τον προπολογισμό, εκτελεί τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να αποφύγουμε εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουμε τον όρο delegated management δηλαδή εξισοδότηση διαχείριση του προπολογισμού, ακριβώ επειδή μπορεί να δημιουργήσει κάποιε παρανοήσει όρο αυτό. Εμεί εκτελούμε, όπω ακριβώ λέγεται και στη συνθήκη, το κοινοτικό προπολογισμό. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποια πιστοδρόμηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά την ανάληψη των ευθυνών της και προφανώς εμεί κάθε φορά θα υποβάλλουμε σε εσά την εκτέλεση του προπολογισμού για να μας δώσετε εσεί απαλλαγή στη συνέχεια. Δεν πρόκειται να γίνονται δημοψηφίσματα τώρα όσον αφορά την εμπλοκή των πολιτών, απλώ θα διαβουλευόμαστε μαζί τους για να δούμε πραγματικά ποια έργα θέλουν να προωθήσουν και στη συνέχεια ερχόμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους εταίρους επιτόπου προκειμένου να ληφθεί και από αυτούς υπόψη η άποψη των Ευρωπαίων πολιτών. Όσον αφορά τώρα τα καταπιστευματικά ταμεία και όσον αφορά την ε, υποβολή των εκθέσεων είναι δύο ζητήματα που θα ήθελα να καλύψω στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου. Um, uh, όσον αφορά αυτό που είπε ο εισηγητής, ότι είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να παρακολουθήσετε την όλη λογική, τη συλλογιστική μάλλον της έκθεσης αυτής, σας υπόσχομαι ότι θα έχετε μία ανάρθρο πλέον παρουσίαση της πρότασης αυτής, με πιο λεπτομερή παρουσίαση της λογικής που διέπει τις διάφορες διατάξεις, όπου θα προβάλλουμε περισσότερο τις πιο σημαντικές διατάξεις της πρότασης αυτής και σε ένα παράρτημα στη συνέχεια θα συμπεριλάβουμε τις λιγότερο σημαντικές δευτερεύουσες διατάξεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε όλες τις πιθανότητες δαπανών, όλες τις μορφές δαπανών και του σχετικού ελέγχου που θα πρέπει να γίνεται για αυτές. Θεωρούμε ότι έχουμε ακολουθήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση και θα ήταν το καλύτερο βέβαια να δούμε ανά κεφάλαιο έπειτα την κάθε πρόταση ξεχωριστά με κάθε δυνατή λεπτομέρεια προκειμένου να διασκεδαστούν οποιασδήποτε ανησυχίες. Πρόεδρος, πολύ ωραία, περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής σας λοιπόν. Ευχαριστώ. Πολλοί έχουν ήδη μιλήσει ευρωβουλευτές για αυτά τα θέματα. Θα έρθω τώρα για μια καλύτερη δυνατότητα διαλειτουργικότητας όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Έχουμε τα δημοτικά ταμεία και άλλα, αλλά όλα αυτά τα μέσα δεν μας διευκολύνουν πάντα να τα συνδυάζουμε. Το ΕΦΣΥ, ευρωπαϊκά μέσα χρηματοδότηση κτλ. Οπότε πρέπει να δούμε πώ θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Τι προτείνουμε, προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε όσα γίνεται περισσότερο ή ενιαίους κανόνες ή κανόνες με συνοχή. Και θα απαντήσω και στις ανησυχίες του κύριου Ολμπριχτ τώρα. Για τα νούμερα. Για να καταλάβετε περισσότερο. Ή που συνδυάζουμε τα χρηματικά μέσα με ε, τα καταπιστεύματα. Γιατί? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Στη μία περίπτωση γνωρίζεις καλά τον ε, εταίρο σου, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις καταπιστεύματα που προβλέπονται για τον οποιοδήποτε. Όταν όμως έχουμε το ΕΦΣΙ με το ESI, τότε προτείνουμε να τροποποιηθούν οι κανόνες των διευθυντικών ταμείων έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδυάζονται με το ESI. Οπότε οι υπόλοιποι κανόνες είναι, ε, έχουν συνοχή με το ΕΦΣΥ. Πρέπει λοιπόν είτε να έχουμε ενιαίους κανόνες είτε να έχουμε κανόνες με συνοχή αλλά όταν μιλάμε για το ESI δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι των χωρών μελών γιατί οι χώρες μέλη λογοδοτούν για αυτά. Συγκεκριμένα για τον συνδυασμό αυτό, για τους ίδιους πόρους. Συνδυασμός ιδιωτικών πόρων, FC και ESI. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τρεις κανόνες. Ένα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα για το ε, Ταμείο Γιούγκερ και το τρίτο για το ESI. Συνεπώς, εδώ τροποποιούμε τους κανόνες ESI, οπότε έτσι δεν υπάρχουν πια τα προβλήματα τα οποία εμποδίζουν τον συνδυασμό του με το EFSI, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, Ταμείο Juncker. Δεν πρόκειται μόνο για ενιαίους κανόνες, γιατί οι χώρες μέλη παραμένουν υπεύθυνοι για τη, χρήση, για τη χρήση, αλλά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις από τους κανόνες CPR που συνδυάζονται με το ΕΦΣΥ για να είναι εφικτή η συνεισφορά αυτή του ΕΦΣΥ, η χρήση των κονδυλίων ΕΦΣΥ. Τώρα ερχόμαστε στην ευελιξία που ήταν η δεύτερη κύρια ανησυχία όπως ο πρόεδρος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ήταν και η κύρια ανησυχία των διαφόρων εταίρων και εδώ έχουμε διάφορες απαντήσεις. Το flexibility cushion για την εξωτερική δράση, έχουμε πιο γρήγορες πληρωμές, έχουμε την άδεια για ευρωπαϊκά καταπιστεύματα προτάσεις που νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα συζητηθούν εκτενέστερα, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πλαίσιο λογοδοσίας και δράσεων στον τομέα των δημοσιονομικών μέσων, των εγγύσεων και της πολυμερούς αρρωγής. Ας δούμε λοιπόν λιγάκι την ευελιξία. Μία πρόταση που έχουμε υποβάλει Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί πρόκειται για εθνικά κονδύλια των ε, διευθυντικών ταμείων, προκειμένου να υπάρχει μεταφορά των κονδυλίων αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την ε, κοινή διαχείριση πηγαίνει στην ε, άμεση έμεση διαχείριση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το αποφασίσουν οι χώρες μέλη. Και θα εφαρμόζονται συγκεκριμένα προγράμματα στην επικράτεια αυτό των χωρών μελών. Παράδειγμα, υπήρχε ένα πρόγραμμα σε, ως εθνικό πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό δεν προχωράει. Η χώρα μέλος ξέρει ότι το πρόγραμμα είναι σε αναμονή για χρηματοδότηση. Είναι για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην επικράτειά του. Αντί να χάσει λοιπόν, αντί να μην χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά, μπορεί να τα μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο κόσμο και να βοηθήσει έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επικράτεια του συγκεκριμένου χώρου κράτους μέλους. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή χρήση αυτή των κονδυλίων που δεχάνουν οι χώρες μέλη. Πάντα για την ε, ευελιξία. Πιο σύντομη διαδικασία. Πρώτον έχουμε την ε, κινητοποίηση της απόφασης και στη συνέχεια έχουμε τον τροποποιημένο κανονισμό. Όλα αυτά παίρνουν πολύ χρόνο. Γι' αυτό θέλουμε να γίνει απλοποίηση και να πούμε ότι άπαξ και υπάρχει κινητοποίηση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης κινητοποιείται για να κάνει τη μεταφορά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Η απόφαση έχει ήδη ληφθεί στο στάδιο της κινητοποίησης. Το ίδιο και για το Ταμείο για τις Επιτώσεις της Παγκοσμιοποίησης. Άπαξ και έχει δοθεί άδεια για την κινητοποίηση, τότε η μεταφορά εγκρίνεται. Όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια με τον τρόπο αυτό φτάνουν πιο γρήγορα εκεί που υπάρχει ανάγκη για αυτά, είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε πρόκειται για κλείσιμο εργοστασίων κλπ. Τώρα, ερχόμαστε στην ευελιξία για τα κατεπιστεύματα. Δεν προτείνουμε με τίποτα αυτά τα trust funds να γίνει η συνήθις πολιτική εφαρμογή της πολιτικής μας. Όχι. Απλώς είδαμε ότι η πρόσφατη μεταναστευτική κρίση έδειξε ότι υπάρχουν όρια στη δράση μας. Δεν είμαστε αποτελεσματικοί αν δεν μπορούμε με μία μεταφορά να καλύψουμε και τις εξωτερικές συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης, αλλά και τις εσωτερικές. Ποιες είναι οι σημερινές συνέπειες μπορούμε να δώσουμε πλήρη στήριξη μέχρι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των και τους μετανάστες. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα, δεν μπορούμε να δώσουμε την ίδια στήριξη. Η κατάσταση είναι περίεργη λοιπόν. Και αυτό που ζητάμε είναι την άδεια να μπορούμε να καλύψουμε και τις εσωτερικές συνέπειες εξωτερικών κρίσεων. Όπως ξέρετε, αν μεταφέρονται τα κονδύλια από τις εσωτερικές πολιτικές σε trust funds, τότε γίνεται. Και υπάρχει φυσικά πλήρης λογοδοσία, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία διαχειρίζεται τα trust funds αυτά. Και έρχεται σε εσά ε, τη στιγμή της απαλλαγής και ενημερώνεστε και έχετε λόγο τότε. Προτείναμε επίσης να αυξήσουμε και τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κατάρτιση, τη δημιουργία των trust funds. Θα πούμε περισσότερα σήμερα το απόγευμα. Έχουμε streamlined reporting για να μην χάνετε πληροφορία. Πρέπει τις πληροφορίες να τις συγκεντρώνουμε με τρόπο που να έχει νόημα σε δύο στιγμές που πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να έχετε τις πληροφορίες. Όλες αυτές οι εκθέσεις λοιπόν συγκεντρώνονται έτσι ώστε να έχουν νόημα και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες και να τις συνδυάσετε με όλα όσα προβλέπονται. Τι προτείνουμε λοιπόν. Τρεις εκθέσεις στο πρώτο επίπεδο που είναι τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνέχεια για τις εκτιμήσεις έχουμε δύο έγγραφα, τώρα θα έχουμε ένα στο μέλλον. Όσον αφορά τώρα την ε, εκθέση για την εφαρμογή, την χρήση του προϋπολογισμού, εδώ δεν νομίζουμε αν αντί να γίνεται και μηνιαία έκθεση και κάθε τρεις μήνες, θα χάσουμε σε πληροφορία αν γίνεται μόνο κάθε μήνα. Και όσον αφορά την ε, ε, επίδοση, επίσης έχουμε βάσει το άρθρο 318. Πιστεύουμε εμείς ότι με μία ενιαία έκθεση είμαστε καλυμμένοι. Για να ολοκληρώσω. Δεν θέλουμε να μειώσουμε την κοινή διαχείριση. Και σαν παράδειγμα της βούλησής μας αυτής ενισχύουμε την προστασία από τις απάτες και τις παρατυπίες αναβαθμίζοντας την καταπολέμηση της φόρα αποφυγής και διευκρινίζουμε και τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για την εισηγήτρια. Τέλος, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σας πείσουμε για το ότι βελτιώνονται οι συνθήκες με την πρόταση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Συμπληρώνει το σύνολο των προτάσεων που είδαμε στο σχέδιο κανονισμού. Η κυρία Γκρέσλε θέλει να μας συνοψίσει τις υπόλοιπες της ε, παρατηρήσεις. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο το θέμα. Ο προσδιορισμός για καταπιστεύματα. Για μένα έχει άλλο νόημα. Ναι, βεβαίω μπορείτε μετά να αρχίσετε να περιορίσετε και τα λοιπά, αλλά παρά είναι ασαφής. Και πάντως δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε πράγματα τα οποία στη συνέχεια δεν θα μπορούμε να ελέγχουμε και να εποπτεύουμε. Πολλά είναι από αυτά τα οποία μας έχετε προτείνει τελείως αδιαφανή. Ο συνδυασμός, σε παραδείγματι, ε, δάνεια και χρηματοοικονομικά μέσα grants και financial instruments. Δεν πρέπει, εφόσον υπάρχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα, να έχουμε την υποχρέωση της, ε, του ελέγχου, της λογοδοσίας. Δεν βλέπουμε με φρίκι μέρα με τη μέρα τόσα προβλήματα στη λογοδοσία ακριβώς στην ε, διαχείριση των πόρων. Δεν μπορούμε λοιπόν να την βγάλουμε μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν μέσα δάνεια. Λέτε ότι η συγχρηματοδότηση διατηρείται, οι όροι, οι κανόνες τη συγχρηματοδότηση. Ναι, οκ. Okay. Και ποιο θα διαπιστώνει ότι όντω τηρούνται στη μεικτή διαχείριση, γιατί δεν θα έχετε κανένα έλεγχο του ποιο κανόνα τηρείται και αν τηρείται οποιοδήποτε κανόνα. Γιατί μπορούμε να έχουμε χιλιάδε κανόνε εδώ και εκεί που θα γίνεται η εκτέλεση του έργου να μην ελέγχει κανεί κανένα κανόνα. Λοιπόν, εγώ αυτά δεν μπορώ να τα δεχθώ με τίποτα Και θέλω πάνω απ' όλα να μπορούμε να διατηρούμε τον έλεγχο του τι γίνεται στην εκτέλεση, στην κάθε περιοχή, στο κάθε σημείο. Απλούστευση, ναι. Αλλά να μην είναι ε, όλο και πιο απλά τα πράγματα μόνο για αυτόν που ξέρει να βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Όπως είπα, βλέπω αρκετά ενδιαφέρουσες, αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις. Ναι, πρέπει να τις βελτιώσουμε. Ναι, πρέπει πάνω απ' όλα να συζητήσουμε, εξάπατος να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο, όπως είπα και νωρίτερα. Ήθελα πιο πολλές πληροφορίες για την άμεση, για την έμεση διαχείριση, πώς εξελίσσονται τα διάφορα στάδια τους, πότε διατίθενται τα ποσά, πότε αποδεσμεύονται, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ότι αυτές οι προτάσεις είναι και εφικτές. Και βεβαίω μακάρι να μπορέσουν να πλουστευτούν τα, τα ποσά έτσι ώστε να μην χάνεται η ουσία της εκτέλεσης. Και μακάρι κάποιοι να πούνε να τώρα θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα ποσά χωρίς προβλήματα. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό το μεγάλο άνοιγμα δεν μπορεί να γίνει με τη λογική ότι έχουμε όλα αυτά τα κονδύλια και επειδή ήμασταν πολύ αυστηροί πριν τώρα χαλαρώνουμε τελείως και δεν κοιτάμε κανένα τι κάνει. Λοιπόν, και όπως είπα, δεν μπορώ να παραιτηθώ εγώ έτσι εύκολα, θα διεκδικήσω εγγυήσει. Έχω και τη γνωμοδότηση εν αναμονή του ελεγκτικού συνεδρίου. Την περιμένω από ώρα σε ώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας δώσει τη δική του την θεώρηση του ελεγκτικού συνέδριου και τις εκθέσεις και τις συστάσεις του. Λυπούμε βαθύτατα που δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Εγώ 19 Μαρτίου καταθέτω έκθεση. Εμείς καταθέτουμε έκθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όχι για να κάνω κανένα στο χατήρι. Πρόεδρος. Δεν έχουμε όμω ιδίου πόρου αυτή τη στιγμή στο κοινοτικό προπολογισμό, άρα όλα τα χρήματα από τα κράτη-μέλη προέρχονται. Άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να ανακτούν ουσιαστικά τα ποσά εκείνα τα οποία εισφέρουν, συνεισφέρουν στο κοινοτικό προπολογισμό. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο όμω να μην παρουσιάζει πολυπλοκότητα. Ο κύριο Άσουορθ, ο συνεισηγητή, θέλει να πάρει το λόγο. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ να θίξω ένα-δύο σημεία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε προφανώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συνειδητοποιούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν, γιατί ακούστηκαν μόνο αρνητικέ επικρίσει. Ενδεχομένω σα μην δοθεί εδώ λανθασμένη εντύπωση. Προφανώς χαιρετίζουμε κάποιες από τις καινοτόμες προτάσεις τους, αλλά χρειάζομαι όμως και εγώ κάποιες διασφαλίσεις, ιδίως για τους ελέγχους. Νέε διαδικασίε μας είπατε πολύ ωραία, αλλά θα πρέπει να μας ικανοποιήσουν και οι νέοι έλεγχοι που προτείνεται. Ένα παράδειγμα. Κατά αποκοπήν ποσά και προτάσει όσον αφορά το κόστος μονάδος. Νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί, μάλλον ακόμα και πέρυσι έκανε μια διαβούλευση με συμμετέχοντες, αν θέλετε, στην πρόταση αυτή με μπλεκόμενα μέρη, οι οποίοι είπαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένη η μέθοδος αυτή. Όσον αφορά τα καταπιστεύματα, δεν καταρρύπτουμε σε καμία περίπτωση την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά τι συστήματα ελέγχου θα έχετε για τα καταπιστεύματα αυτά. Αυτό περιμένουμε να μας πείτε. Και κάποιες αβεβαιότητες, αμφιβολίες εξακολουθούν και υπάρχουν σε σχέση με το ΕΦΣΥ και σε σχέση με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα. Θυμάμαι ότι την εποχή του ΕΦΣΥ είχαμε πει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν μία επέκταση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και παιδιτικών Ταμείων. Υποτίθεται ότι το ΕΦΣΥ θα αντιμετώπιζε νέε προκλήσει νέα γενιά, καθώ επίση και επενδύσει νέα γενιά, όπω μα είχατε πει τότε. Και τώρα τι βλέπουμε. Έρχεστε και παρουσιάζετε το ΕΦΣΥ ω μια απλή επέκταση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση το ΕΦΣΥ, το οποίο παρουσιάστηκε ως πρωτοβουλίο ορόσημο για νέες επενδύσεις, να αποδυναμωθεί και να αποτελέσει απλώς ένα τμήμα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Σας ευχαριστώ πολύ αυτές την παρατηρήσεις μου και ελπίζω πραγματικά να επωφελήσει ναι, αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Πυρίνσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι και εγώ σύντομος. Πρώτον, όσον αφορά τη διαφορά ημί μεταξύ Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και ΕΦΣΥ, καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την όλη συλλογιστική που μας εξέθεσε πριν από λίγο, ότι δηλαδή οι κανόνες για τα διαφορετικά ταμεία θα πρέπει να προσαρμοστούν στους κανόνες για το ΕΦΣΥ, γιατί αυτό απαιτεί, μας είπατε, η αγορά. Μα όπως το είπατε κι εσείς, ο προπολογισμός προϋποθέτει, προβλέπει μια ανακατανομή πόρων και σε καμία περίπτωση, και ιδίω όσον αφορά το τμήμα τη συνοχή, δεν εξυπηρετεί, δεν θα πρέπει να εξυπηρετεί την αγορά. Εξυπηρετεί τον ε, απότερο στόχο της συνοχής, της μείωσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, της μείωσης των οικονομικών, κοινωνικών διαφορών, αποστάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ κρατών μελών. Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να λέτε ότι όλοι όλα αυτά τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία τα οποία προγραμματίζουμε εμείς πώς θα χρησιμοποιηθούν σε πολιετή βάση, ότι ξαφνικά θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το οποίο μας είπε μόλις τώρα ο κύριος Ashworth, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου ανά πρόγραμμα. Αυτό είναι παράλογο και δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει λόγος να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όσον αφορά τώρα το σύστημα διαχείριση, καθώ επίση και την εκτέλεση του προπολογισμού, μα είπατε αυτή τη στιγμή ότι η συνθήκη μιλάει για implementation στα αγγλικά και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε τον όρο αυτό και εσεί. Αλλά από την άλλη, μα είπατε αυτή τη στιγμή πάρα πολλέ φορέ χρησιμοποίησατε άλλου όρου. Μα είπατε ότι μιλάτε για management, αντί να μιλάτε για implementation. Μιλάτε για διαχείριση του προπολογισμού και όχι για εκτέλεση προπολογισμού στην πρότασή σας. Μήπως λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μιλάτε περισσότερο για χρηστή εκτέλεση του προπολογισμού και όχι τόσο πολύ για χρηστή διαχείριση του προπολογισμού όπως κάνετε σε πάρα πολλά σημεία της πρότασής σας. Για τα καταπιστευματικά ταμεία μας είπατε ότι είναι τμήμα πλέον του προπολογισμού και αυτά και ότι στο παράρτημα 3 λέγεται ότι μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τα ταμεία αυτά, διαχωρίζονται σαφώς από τον κοινοτικό προπολογισμό ή από ε, βασικά παγιωμένα ταμεία του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μας είπατε ότι τα καταπιστευματικά ταμεία, τουλάχιστον αυτό διαβάζω στο παράρτημα, δημιουργούνται, θεσπίζονται μέσω συμβάσεων που γράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους εταίρους. Αν πρέπει λοιπόν να ζήσουμε στο μέλλον με καταπιστευματικά ταμεία, τότε ας δούμε από πού ακριβώς χρηματοδοτούνται. Εγώ βλέπω ότι έχουν αρχίσει να παίρνουν χρήματα από άλλα παγιωμένα προγράμματα. Αν πάρει το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική, το συνολικό ποσό είναι 1 δισεκατομμύριο 980 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ο κοινοτικό προπολογισμό έχει δώσει 1 δισεκατομμύριο 899 εκατομμύρια, με συγχωρείτε. Και το υπόλοιπο ποσό έχει προέλθει από άλλους πόρους. Επομένως, ουσιαστικά τι λέμε αυτή τη στιγμή ότι προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε ως το δυνατόν περισσότερα χρήματα από ένα κοινοτικό προπολογισμό που ήδη είναι αρκετά περιορισμένος και ουσιαστικά φερώντας χρήματα από άλλα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να πληκοδοτούνται από τον ίδιο τον κοινοτικό προπολογισμό. Euh, Ευχαριστούμε, κύριε Σόλμπριχτ. Ακριβώς μετά από αυτά που είπε ο προλαλής σας, δεν είναι ότι είναι παράλογο είναι ότι έτσι γίνεται και δεν γίνεται τυχαία. Αυτή είναι η λογική του συστήματος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Πώς θα αλλάξει ο ίδιος ο χαρακτήρας χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ζητάμε τεχνικά. Ζητάμε την αλλαγή φιλοσοφίας. Μεταφέρουμε τα χρήματα από τον προπολογισμό σε άλλα μέσα αλλάζουμε την ε, χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική και αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα το απόγευμα. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Συμφωνώ με από την αρχή το ΕΦΣΥ ήταν εντελώς διαφορετικό από τα αρχιτεκτονικά ταμεία. Ήταν πράγματι για προγράμματα υψηλού κινδύνου. Αν τώρα, και είναι αλήθεια, και θα υπογράψω πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι παρατηρήσει τη επιτροπή. Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει για το επενδυτικό ταμείο, για το ΕΦΣΥ και διαφορετικά για τα διαφορετικά ταμεία, διαφορετικές προϋποθέσεις. Αλλά υπάρχει τάση να μεταφέρουμε τα προγράμματα από τα διαφορετικά ταμεία στο επενδυτικό ταμείο, στο ΕΦΣΥ, όπως κατασκευή ε, οδοπίας να πάει από τα ιδιωτικά ταμεία στο ΕΦΣΥ. Αυτό που προτείνει τώρα όμως λέει να μεταφέρουμε τα χρήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καλά στα διευθυντικά ταμεία να πάνε στο ΕΦΣΥ. Αυτό θα είναι προσωρινό ή μόνιμο. Θέλουμε να αλλάξουμε τη δομή του προπολογισμού ή θέλουμε προσωρινά να βρούμε μια στρατηγική εξόδου αφού δεν γίνεται να εξοδευτούν τα χρήματα εκεί, ας πάνε στο ΕΦΣΙ, εκεί θα εξοδευτούν πιο γρήγορα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο τέτοιο οργανισμό. Ίσως να μην το κατάλαβα καλά, αλλά είναι κάτι που για μένα θυμίζει αυτό, στρατηγική εξόδου. Πρόεδρος. Ξέρετε πώς δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών ε, Επενδύσεων. Ήρθε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. και διαπίστωσε ότι 10 χρόνια δεν έχουμε αρκετές επενδύσεις, οπότε και αφού δεν υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό, δημιουργούμε ένα μέσο οικονομικής μόχλευσης. Είναι καθαρά δημοσιονομική μηχανική δεν πειράζουμε καθόλου το τμήμα των χωρών μελών. Όταν φτιάχνουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, βάζουμε 80% στην πάντα για την κοινή γεωργική πολιτική και για τα διαρθρωτικά ταμεία, ταμεία συνοχής. Και δεν τα πειράζουμε αυτά, γιατί κάθε χώρα θα πάρει το δικό της κομμάτι και κάθε χώρα πρέπει να επαληθεύει ότι έχει όντως πάρει, έχει πάρει πίσω τα χρήματά της. Συνεπώς, πήγαμε να βρούμε χρήματα σε κάτι που είναι υπερεθνικό. Ορίζοντας 2020, διευκόλυνση για την Ευρώπη, για να βάλουμε λίγα χρήματα στον κουμπαρά, ώστε να μπορέσουμε 21 δισεκατομμύρια, 5 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 6 από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, επί 3,63 και είπαμε, όσοι δανειστείτε πρέπει να τα προσθέσετε επί 5 για να μπορέσετε να αποφεληθείτε με την απλοποίηση. Μερικές φορές ασχολούμαστε με περιθωριακές περιπτώσεις και στο δικό μου το τμήμα το είχα ένας πρόεδρος Επιτροπής Δημοποίησης ζήτησε κάποια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπα μάλιστα ναι υπάρχει το πρόγραμμα για τους Ευρωπαίους πολίτες λοιπόν πήρε το φάκελο 50 ώρες να το συμπληρώσει, το πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του είπανε μάλιστα αξιολογήσαμε, πήρατε 50% αλλά χάσατε γιατί έπρεπε να έχετε πάρει 76% για να πάρετε επιδοτήσεις. Για μερικέ. χιλιάδες ευρώ έχει νόημα να δημιουργούμε τέτοια απογοήτευση ή δίνουμε λίγα χρήματα χωρίς να το ψάχνουμε πολύ για το αν πληρώσανε κοκακόλα 12 ευρώ ή 10 ευρώ το μπουκάλι. Δηλαδή Πρέπει να ξέρουμε αν θέλουμε να παρεύουμε ή δεν θέλουμε να παρεύουμε. Αν υπάρχει επικουρικότητα, υπάρχουν και πράγματα που είναι περισσότερο αρμοδιότητα των χωρών μελών από ό,τι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δημιουργεί γραφειοκρατία, απασχολεί κόσμο, υπηρεσίε και δίνει και μια πολύ άσχημη εικόνα τη Ευρώπη. Φανταστείτε αυτό ο Δήμαρχο που ήθελε τη δημοποίηση, τι θα εξηγήσει στου πολίτε του όταν κάθισε και πέρασε 50 ώρε να συμπληρώσει το φάκελο και μετά του είπανε Α, δεν θα πάρετε τίποτα. Λοιπόν, ή που θα το κάνουμε ή που δεν θα το κάνουμε. Καλύτερα μερικέ φορέ να μην το κάνουμε καθόλου. Είναι ήδη περίπλοκα τα πράγματα για τις περιφερειακές τράπεζες να ασχολούνται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φανταστείτε να πρέπει να είναι στις Βρυξέλλες που θα ασχολούνται με αυτό. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα, ακόμα και αυτά που είναι θέμα επικουρικότητας. Προσοχή! Γιατί η Ευρώπη δημιουργεί προσδοκίες που δεν μπορεί να ικανοποιήσει ή τις εικονοποιεί με τόσο μεγάλο γραφειοκρατικό έλεγχο, κομισιών, υπηρεσίες, τα λοιπά που είναι φρίκη. τα μικρά προγράμματα είναι αυτά που μας δημιουργούν ε, πρόβλημα. Ή πρέπει να τα κάνουμε με ένα κατακοπή κόστος, και τελείως η έλεγχη είναι τόσο μεγάλη και το περιθώριο σφάλματος δεν είναι τόσο... Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το έργο σας πολύ σημαντικό. Τώρα όμως μένει πολλή δουλειά ακόμα και για σας και για μας. Εσείς έχετε την τάση, καταλαβαίνω, να πείτε εμείς τα κάναμε, κορσέ, αλλά δεν πρόκειται να βγούμε έτσι από το πρόβλημα. Να απλοποιήσουμε, να απλοποιήσουμε. Πόσες σελίδες? 780 σελίδες. Μα, αυτό δεν έχει νόημα. Σε 10 σελίδες θέλουμε κανονισμό. Είναι όπως οι εκθέσεις που φτιάχνουμε εμείς, ο κύριος Μπέκε και η κυρία Μπέρες, θα ετοιμάσουν έκθεση σε τρει σελίδε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Συχνά όμω οι εκθέσει μα εδώ είναι 40-50 σελίδε. Κανένας δεν μπορεί να τα διαβάσει. Αδιαφορεί ο κόσμος. Δεν τα διαβάζει. Είναι απλώς για να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, εκεί είναι που πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία στην προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Τι δυνατότητα έχουμε να μιλήσουμε στους πολίτες. Γιατί όταν μιλάμε στους πολίτες, εκείνοι θα πιέσουν τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι βέβαια είναι πάντα με δεμένα τα χέρια, γιατί όλοι και κάποια εκλογή θα έχουν μπροστά τους και έτσι η Ευρώπη είναι στάσιμη. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο ήμιση της θητείας μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Βαλουρόη, λοιπόν, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν ε, πρόκειται να κάνω νέα ανάλυση. Θέλω μόνο να απαντήσω στις τελευταίες παρεμβάσεις για τους πυρογνώμονες και τον κίνδυνο. Τους επιλέγουμε με τις ίδιες προϋποθέσεις που ε, επιλέγουμε και τους ειδικού για την έρευνα. Δηλαδή κοιτούμε να δούμε τι παραγματογνωμοσύνη έχουν. Κάνουμε επιλογή με διαφάνεια. Και σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ανησυχούμε για κάποιο κίνδυνο. Για το έτσι. Πολύ σημαντική παρατήρηση και βέβαια για τους αδέλφους που μεταφέρουν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα εθνικά προγράμματα για το κόσμο, παραδείγμα, σας έδωσα ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε ανοιχτές πόρτες ε, να παραβιάσουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν λέμε ότι ε, θέλουμε να ε, πάρουμε τους πόρους από τα διαφορετικά ταμεία. Αλλά θέλουμε να υπάρχουν οι δυνατότητες, αυτές οι δύο δυνατότητες που αναφέρουμε, θα ισχύουν μόνο εάν αποφασίσει το κράτος μέλος να τα αντλήσει τα ποσά από το έτσι, μέσω, για το έτσι μάλλον, από το εθνικό του πακέτο. Δεν προτείνουμε δηλαδή τίποτε. Δεν προτείνουμε δηλαδή κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι τομείς και αυτή είναι οι αυτές εθνικές πλατφόρμες που θα το προσδιορίζουν και που θα το δώσουν το αποτέλεσμα ότι μπορεί το έτσι να συνδυαστεί με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και μόνο σε αυτήν την περίπτωση, όταν δηλαδή φανεί ότι μπορεί να υπάρχει ένα δυναμικό, μια δυνατότητα για ε, καλά αποτελέσματα στο κάθε κράτος μέρος, Ας μην το καταδικάσουμε. Καταπιστεύματα. Δεν σας είπα εγώ νομίζω ότι είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, σας είπα και το επαναλαμβάνω ότι η εσωτερική λογιστική έλεγχη, η λογιστική, η τήρηση των βιβλίων δηλαδή και οι ευθύνε τη Λογιστική Επιτροπή παραμένουν απαράλλακτοι. Παραμένει η ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η λογοδοσία εναντί ημών για την εκτέλεση των σχετικών λογαριασμών και αυτό θα συμβεί. Ανησυχίε για κονδύλια που προέρχονται από κοινοτικά προγράμματα και μπαίνουν σε καταπιστεύματα βεβαίω υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει είμαστε στη διάθεση σας για να συνεργαστούμε για περαιτέρω οργάνωση των διευθυντικών ταμείων των καταπιστευματικών, των καταπιστευμάτων, συγγνώμη. Ε, ιδιαίτερα για τις Τουρκία θα έχουμε τη συζήτηση και σήμερα το απόγευμα. Ο, το, ο στόχος πάντως είναι στο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα, μεγαλύτερη μόχλευση δηλαδή από τα κονδυλία που ε, διατίθενται. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Και την επιρροή τους δείκτες επιρροής που τους αντλείτε. Πώς αντιμετράτε την επιρροή. Ή η Πρόεδρος. Και συν... Κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, ιδιαίτερα του συναδέλφου με όλες τις προτάσεις και τις ιδέες που μου προσέφεραν. Δεν ήταν ξεκάθαρο το πώς θα διαμορφώνονταν οι θέσεις σας προκαταβολικά. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Άλλο τίποτα επί της ουσίας δεν θα προσθέσω. 19 Μαρτίου θα δείτε την έκθεση, αλλά όπως είπα κάθε ευκαιρία και συζήτηση είναι ευπρόζεκτη. Σήμερα ήταν σημαντικό ότι μπορέσαμε να δούμε ότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία μπορούμε να πάρουμε κάποιε εξηγήσει. Χρειαζόμαστε ακόμα διευκρινήσει. Θα κάνουμε το εργαστήριο εκείνο με το οποίο θα συζητήσουμε και κάποια σημαντικά ε, θέματα. Και βεβαίω όλοι οι συναδελφοί είναι προσκεκλημένοι και από την Επιτροπή των Προπολογισμών και από τον έλεγχο. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ευκαιρία και βέβαια παραμένουμε σε επαφή. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Κύριε Άσχουρθ. Όχι. Ωραία. Πολύ επικοδομητική η πρόκληση στην οποία αποδιόμεθα με πολύ έντονο πολιτικό χαρακτήρα και επιμένω, κατά κύριο λόγο πολιτικό. Και πρέπει έτσι και εμείς να ξέρουμε και τι θέλουμε. Πρέπει να μπορούμε να εξετάσουμε κάθε λύση. Πρέπει να μπορούμε να δείξουμε ε, πειθαρχία, πνεύμα πειθαρχημένο. Και βέβαια ταυτόχρονα να είμαστε και να αναλάβουμε κίνδυνου, κινδύνους, γιατί χωρίς κινδύνους δεν γίνεται δουλειά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ευτυχία για τον καθένα και την καθημεία από σας για το 2017. Κυρίσω την διακοπή της συνεδρίασης για να ξαναρχίσουμε στις 3 με το εργαστήριο για το δημοσιονομικό στερέωμα.